Good afternoon, colleagues. We will start our meeting. Γεια σας συνάδελφοι. Καλησπέρα και αρχίζουμε την ε, συνάντησή μας. Το πρώτο μας ε, θέμα στη μέση διαδέξη είναι η έγκριση αυτή και θέλω να σας πω ότι στο 10 για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας για το 18 το θέμα αυτό έχει αναβληθεί και θα πάει στις 6 ε, ενδεκάτου, ενεστώτος έτους. Ε, αν δεν έχουμε κάποια άλλη ένσταση η παρατήρηση εγκρίνεται η μέση διάταξη και το επόμενο τώρα ζήτημα είναι το υπαριθμόν 2, οι ανακοινώσει τη Προέδρου. Το 2-1. Έχουμε τη συνάντηση τη Τετάρτη Ενάτου των Συντονιστών που απεφάσισαν να δοθεί η έκθεση για τις γυναίκες ως ε, ε παράγοντα τη διαμόρφωση των εξελίξεων στο, ε, στους και επίσης είπαμε ότι οι γυναίκες ως φορείς αλλαγής στις χώρες ε, εταιρική σχέσης με του Νότου και συναφή θέματα. Επίσης έχουμε την μέρα της γυναίκας του 2018 για γυναίκες και νεαρές γυναίκες ως ε, κλειδί για το μέλλον. Έχουμε επομένως τρία εργαστήρια για την μέρα αυτή της ε, γυναίκας, για την χειραφέση της ε, γυναίκας, για την είσοδο στην ψηφιακή εποχή και όπως είπαμε στις 13 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν οι συντονιστές να οργανωθούν οι εξής αποστολές για το πρώτο εξάμεινο του 18 Ουγγαρία τον Φεβρουάριο, Σουηδία τον Μάιο και Ρουμανία τον Μάιο. Και είπαμε ότι θα υπάρξει και το Policy Department ένα σχετικό γραφό για τι γυναίκε ω παρελαγέ επίση. Έχουμε αυτή την αντιπροσωπεία για τι σχέσει με το ε, Ισραήλ. Οπότε σα ε, ενημερώνουμε ότι η ανταλλαγή των απόψεων με την Επιτροπή όσον αφορά την κατάσταση της γυναίκας και την ισότητα του Ισραηλινού Κοινοβουλίου οργανώθηκε από το αντιπροσωπεία μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ για τις 27 Ενδεκάτου του 2017. 5 με 6,5. Και είμαστε όλοι προσκεκλημένοι να λάβουμε μέρος αυτή την συνάντηση. Τελευταία δε ανακοίνωση σας ενημέρω για το εξής. θα υπάρξει κάποια κινηματογράφηση στην συνάντηση. Ε, κατά έτσι της κυρίας Βετλάνσκα. Πάμε παρακάτω τώρα στο σημείο υπαριθμών 3, έγκριση των πρακτικών της 26ης έκτου. Αν δεν έχετε παρατηρήσει η ένσταση, εγκρίνονται αυτά τα πρακτικά. Τέσσερα. κοινοεργαστήριο όσον αφορά τον μετασχηματισμό της ζωής γυναικών και νερών γυναικών η σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλώ ορίσατε στη σημερινή συνάντηση που την οργανώνει το Policy Department για τα δικαιώματα των πολιτών και έχουν σχέση με το πώς θα αλλάξει επομένω μέσω των εξωτερικών σχέσεων η ζωή γυναικών και νεαρών γυναικών. Έχουμε συμπρόεδρο τον κύριο Πόγκα, τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΔΕΒΕ που συνεργώνει αυτή τη συνάντηση. Αντικαθιστά την κυρία Μάκαβαν, η οποία είναι και συνεισηγήτρια για το θέμα μας αυτό. Και μετά αυτό το εργαστήριο έχει συνάντηση η Επιτροπή ΔΕΒΕ και εμείς όμως. Και ευχαριστούμε. Ε, κύριε Πόγκα, έχετε τον λόγο για να μας ε, ενημερώσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να καλωσορίσουμε όλοι κάποιους προσκεκλημένους, οποίους εγώ προσεκάλεσα και πρόκειται για επισκέπτες από το Παρίσι. Οπότε από πλευράς μας, από πλευράς α, Επιτροπής ε, Ανάπτυξης και ε, θεμάτων ε, που αφορούν τις γυναίκες, καλώς ορίσατε φίλοι από το Παρίσι. Η πρόεδρος θωρώνοντα τα πλαίσια τη προετοιμασία τη κοινή έκθεση των όσον αφορά το έγγραφο το κοινό, όσον αφορά την ε, αλλαγή στι γυναίκε νεαρών και νεαρών γυναικών. Ε, καλούμε συζήτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Υπηρεσία Ειδική ε, Δράση σύμφωνα με το έγγραφο τη 21 η Ενάτου του 2017 και οι συνεισηγητές της έκθεσης, η κυρία Σουίτσα και η κυρία Μάκαλαν. Είναι αυτές και πάντως θα πρέπει να ευχηθούμε καλώς όρισαν και οι εμπειρογνωμονές μας οι οποίοι έχουν προσκληθεί για να μας βοηθήσουν να εξετάσουμε τις διάφορες πτυχές ε, της εξωτερικής δράσης ε, που αφορούν ε, τα θέματα των ε, γυναικών. Για να δώσουν τώρα τον λόγο. Στον κύριο Τζιν Λόις Βίλα, τον ε, διευθυντή της ΔΕΒΚΟ. Έχετε πέντε λεπτά κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πρόκληση περισσότερο για τους διερμηνείς ότι έχω χιλιάδες πράγματα να πω και ίσως θα μιλάω γρήγορα οπότε αν δεν με ακούτε κάντε μου ένα νόημα αλλιώς δεν θα σταματήσω πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ θα προσπαθήσω να μοιραστώ την παρουσίαση με την κυρία Μαρινάκη από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι κοινή προσπάθεια, κοινά λοιπόν τα έγγραφα, τα οποία βλέπετε ε, λίγα λόγια. Πάρα πολλά κάτι όχι τόσο σημαντικό, αλλά σημαντικό κάπως. Ο ΙΕ και τα κράτη-μέλη βεβαίως προωθούν την ισότητα των φίλων και την ενδυνάμωση των γυναικών σε εξωτερικές σχέσεις και αυτό φαίνεται στην έκθεση αυτή και είναι προφανές αλλά μια φορά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε αυτά η έκθεση αυτή λοιπόν συντάσσεται για πρώτη φορά μετά την έγκριση του πενταετούς σχεδίου. Είναι υποχρεωτικό για όλες τις αντιπροσωπείες της Ένωσης. Έχουμε λάβει 108 απαντήσεις από τις αντιπροσωπείες ε, που καλύπτουν περίπου το 80% της επιφάνειας ε, της Ιφιλίου. 133 χώρες δηλαδή, καθώς ε, κάποιες αντιπροσωπείες καλύπτουν περισσότερες χώρες. Συνολικά, 26 αντιπροσωπείες δεν ε, υπέβαλαν αναφορά, έχουν σοβαρούς λόγους. Κάποιοι γιατί η χώρα την οποία καλύπτουν ε, βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση όπως η Συρία. Σε άλλες περιπτώσεις είναι αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΩΣΑ, οπότε δεν έχει αντικείμενο. Τέσσερις λοιπόν προτεραιότητες είχε η έκθεση. Θα προσπαθήσω έτσι να τα διατρέξω κάπως γρήγορα. Και να εστιαστώ στην πρόοδο του 2016. Λοιπόν, έχουμε έναν στόχο να ενσωματωθεί η δράση του φίλου στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας μέχρι το 85% τουλάχιστον. Ε, πολύ δύσκολο αυτό βεβαίως, γιατί σημαίνει πως έχουμε η διάσταση του φύλου ε, στο 85% των προγραμμάτων μας. Ε, τα αποτελέσματα για το 2016 είναι στο 58,8% σχεδόν 60% των νέων δράσεων είναι προσανατολισμένες ή ευαισθητοποιημένες για το φύλλο σύμφωνα με την ονοματολογία που χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Για τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ κονδυλίων, κάτι το είναι αρκετά καλό. Όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφέ, γιατί ζητούσαμε από τι αντιπροσωπείε μα να κάνουν έναν αριθμό δράσεων. Υπήρχαν πέντε σημαντικές. Πρώτα απ' όλα δηλαδή η χρήση ή η δικαιολόγηση μια δράση που δεν είχε διάσταση του φίλου και έπρεπε να εξηγήσουν γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, οπότε πρέπει να γίνεται αυτή η ανάλυση. Δεύτερον, να γίνει μια ανάλυση του φίλου στην χώρα και εκεί πέρα είχαμε αρκετά καλά αποτέλεσμα γιατί είχαμε 46 αναλύσεις που ενημερώθηκαν οι συνετάξεις μετά να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα αναλυμένα για να ξέρουμε τι και πώς επηρεάζεται ε, γιατί χωρίς αυτό δεν ξέρουμε τι γίνεται και είναι δύσκολο μετά βεβαίως να προσανατολιστούμε στο τι θα κάνουμε και ε, βεβαίως ε, να υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη φίλου είτε μέσω κάποιου ειδικού στην αντιπροσωπεία είτε μέσω εξωτερικής στήριξης και βεβαίως ε, στόχος να υποστηρίζεται από το σχέδιο δράσης. Αυτά είναι τα πέντε πράγματα. Από τις 108 εκθέσεις ήδη 11 ε, προσωπίες είχαν 5 παραγραφές και μετά κάποιες άλλες 4, 3 και τα λοιπά. 7 αντιπροσωπείες δεν ε, πλήρωσαν κανέ, καμία από τις 5 παραγραφές, κάτι το οποίο ε, είναι βεβαίως δυσάρεστο, αλλά 7 είναι και μικρός αριθμός. Μετά η έκθεση, του σχέδιο δράσης, με συγχωρείτε. Από έφτασα τα 5 λεπτά ήδη. Το σχέδιο δράσης εστίασε σε τρεις θεματικές προτεραιότητες και μία για μια πολιτισμική αλλαγή και θεσμική αλλαγή. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία επέλεξε να πάει στο θέμα της σωματικής και ψυχολογικής ακαιρεότητας, το πιο προφανές, δηλαδή μιλάμε για βία κατά των γυναικών, Το δεύτερο βεβαίω είναι η οικονομική ενδυνάμωση και το τρίτο η πολιτική συμμετοχή. Για το μέλλον τώρα, για θα προσπαθήσω να συντομεύω, χρειαζόμαστε. Ε, μια σύσταση δηλαδή που έχουμε κάνει είναι... Να, έχουμε χρόνο, μάλιστα, μάλιστα. Ε, τότε να μιλήσω άλλα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο. Δεν θα σας εξηγήσω βεβαίως, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να εμφυλιωθεί πολύ περισσότερο. Πρόκειται λοιπόν για μια κατεύθυνση προς την οποία θα θέλαμε να πάμε. Δεύτερον, θέλουμε να προωθήσουμε την εφαρμογή αυτή των στόχων ε, μέσω του προσωπικού, όχι βεβαίω μέσω μόνο των ατόμων των υπευθύνων, αλλά να πείσουμε τα υψηλότερα κλιμάκια των επικεφαλής αντιπροσωπείας, των επικεφαλής συνεργασίας, αλλά και στα κεντρικά. Έχουμε μία επίτροπο και ένα γενικό διευθυντή που είναι βεβαίω πολύ υπέρ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι σε όλα τα επίπεδα ε, ανταποκρίνονται 100%. Βεβαίω, ε, επιμένουμε στο ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή, όχι μόνο αρμόδιος και ε, η Επίτροπος. Και οι δύο είναι αναγκαίοι, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Ολόκληρη η δομή πρέπει να ασχοληθεί με την διάσταση του φύλου για να έχουμε αποτελέσματα. Λοιπόν, νομίζω, έχω λίγο χρόνο. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω τον λόγο στην Μαρία, αν μου επιτρέπετε. Thank you very much. Yes, please. Uh, now Ambassador Mara Marinaki, please. Thank you, thank you, Chair. Κυρία Μαρινάκη, ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ζων Λουί διότι ήταν εξαιρετικές εισαγωγικέ του παρατηρήσεις και καλέ αναφετηρία και έχουμε αυτή την πρώτη εφαρμοστική έκθεση για αυτό το πρόγραμμα. Αυτά μας βοήθησαν στις προσπάθειές μας να έχουμε ένα όχημα πρόοδου ούτως ώστε να αλλάξουμε, να μετασχηματίσουμε την αλληλεγγύη των γυναικών και των νέων γυναικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εξωτερικής δράσης. Και θα πρέπει να έχουμε στοχευμένες προσπάθειες ούτω ώστε να χειραφετηθούν οι γυναίκες και να πετύχουμε την ισότητα. Οπότε έχουμε εδώ ένα πολύ εύστοχο μείγμα των αρίστων πρακτικών και των επιτευγμάτων. Οπότε και θα πρέπει να εστιάσουμε προσευχές μας στο πώς θα βελτιώσουμε περαιτέρω τα πράγματα είναι αυτονόητο ότι ήδη κινητοποιηθήκαμε, ήδη βελτιώσαμε την κινητοποίησή μας για όλες τις 140 αντιπροσωπείες μας παγκοσμίω. Και επίσης όλα τα σημεία δράσης της εξωτερικής δράσης και έχουμε ήδη προσπαθούμε να καλύψουμε την ισότητα των νέων, να καταπολεμηθεί η βία, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει ώστε να αλλάξει η ζωή γυναικών και νεαρών γυναικών. Δεν μπορούμε να έχουμε βελτιώσεις εάν δεν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Θα πρέπει να αισθάνονται χειραφετημένες οι γυναίκες, αλλά πρώτα να αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά την ίδια τη ζωή τους. Οπότε είναι κοινή προσπάθεια αυτή με τον ΟΗΕ. αυτόν τον το που θέλουμε από κοινού να στείλουμε. Έτσι και έγινε πρόσφατα και ξεκίνησε με αυτή την πρωτοπόρα κοινή πρωτοβουλία που ονομάζεται Spotlight. Ξεκίνησε πριν από τρει μέρες. Είναι η κοινή μεταξύ του, του Γενικού Γραμματέα του κ. Μοχάμεθ, της κυρίας Μογκερίνη και του Επιτρόπου Μίμιζα που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την πρωτοβουλία, ούτω ώστε να εξαλείψουμε την κατά των γυναικών βία παγκοσμίω. Τώρα, επίσης αυτό το κάνουμε και θα υλοποιήσουμε την ευαισθησία μας σε σχέση με το θέμα του 2030 κανείς να μην μείνει απ' έξω και έτσι να εντάσσουμε αυτή την προσπάθεια στους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης και θέλουμε να υπάρχει τέτοιου είδους ε, ανθρωπιστικός δεσμός ας πούμε του, ε, της μιας με την άλλη υπέρ των γυναικών συγκρούσεις βία να καταπονομηθούν, ισότητα να προωθηθεί στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών και μέσω των φορέων των γυναικών και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα έχει προτεραιότητα ούτως ώστε να προστατεύσουμε ουσιαστικά τις γυναίκες και επίσης να υπάρξει feedback από τις γυναίκες και να καταφέρουμε οι πολιτικές μας να έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή. Να βοηθήσουμε ε, επίσης τους αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κάνουν προσπάθεια παντού και έτσι να υλοποιήσουμε την δέσμευσή μας για το θεμετόλο 2030. Να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, αλλά βεβαίω και υπολογίζουμε στην προσπάθεια του Ευρωπαϊκού, τη βοήθεια μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κυρία Μαρινάκη, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα. It's okay for you to sit here? No? It's okay to sit? It's not? You're not safe? <laughs> okay. Okay. Uh, okay, and now I'd like to give the floor to... Uh, uh το λόγο στον ε, δόκτωρα Πέτρεσεν από το Δανέζικο Ίδρυμα Διεθνών Σπουδών. Έχετε το λόγο, κυρία Πέτρεσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκλησή σας να έρθω να σας μιλήσω για αυτά τα θέματα να σας πω για την ισότητα των δύο φίλων για τη χειραφέτηση των γυναικών, ιδίω όσον αφορά την Αφρική, όσον αφορά επίσης ε, την πολιτική πλευρά του θέματος. Αυτό είναι στόχος φιλόδοξος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπει κανείς παντού όπου υπάρχει αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό είναι και το θέμα. Πρώτα-πρώτα να σας πω στη συγκυρία στην οποία κινούμεθα θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι αυτοί οι κανόνες, οι στόχοι αλλάζουν μέσα χρόνο. Δεν είναι κάτι διαχρονικό, ούτε είναι και κάτι όμως που πάντοτε λαμβάνεται υπόψη. Και είπαμε ότι υπήρχε ενθουσιασμός τέλος δεκαετίας του 90 ήταν πολύ σημαντικό ως ε, θέμα, ως υπόθεση, αλλά τώρα γίνει στροφή. Ε, για περισσότερο προσανατολισμό προς το ίδιο θέμα. Πάντως και το περιεχόμενο της προσπάθειας έχει αλλάξει. Η χειραφέτηση ε, τώρα έχει περισσότερη οικονομική χρειά. Αυτό το προστίζει και η Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι ξεκίνησε σε σχέση με κάποιες διαφορετικές αλλαγές που αφορούσαν τις ε, συνθήκες ε, ζωής των γυναικών. Οπότε όλα αυτά σημαίνουν ότι το σκηνικό έχει αλλάξει και αλλάζει συνέχεια. Επίσης έχουμε ασχοληθεί σε, με ένα ερευνητικό πρόγραμμα όσον αφορά το πώς ε, Αυτέ οι προσπάθειε το Ίδρυμα Gates, η Oxfam και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν βοηθήσει αυτή την υπόθεση και καταλήξαμε στο ότι η οργανωτική προέλευση αυτών των ε, φορέων επηρεάζει την προσπάθεια για επίτευξη ισότητας. Έχει γίνει επομένως μια τέτοια στροφή. Πρέπει να ληφθεί η υπόψη επίσης και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι προκλήσεις αφορούν την χειραφέτηση και την ισότητα και είναι σημαντικός ο ρόλος πολλών φορέων. Αλλά υπάρχουν πιέσεις, υπάρχει η κάθε εθνική πολιτική που επηρεάζει τις προτεραιότητες. Ε, και επίση έχει σημασία το τι γίνεται σε κάθε κέντρο αποφάσεων. Τώρα, όσον αφορά τι αλλαγέ σε επίπεδο κάθε χώρας, έχουμε τι προτεραιότητε οι οποίε μεταβάλλονται. Είναι πολλέ. Πολλέ φορέ υπάρχει πρόβλημα προσωπικού. Πολλέ φορές ε, μερικά απασχολούμενοι, νεότεροι από τους εργαζόμενου σε αυτό το μέτωπο και έτσι δεν μπορούμε να καλυφθούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε το κατάλληλο περιθώριο ελιγμών. Σε κάποια κοινωνικά συστήματα δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Επομένω, αυτό δεν βοηθάει την υπόθεση του θεματολόγιου σαν συμπέρασμα. Να πούμε ότι πολλέ αυτέ, πολλέ φορέ, ε, είναι κάτι, μια, μια τυπικότητα αυτή η προσπάθεια για την ισότητα. Δεν βοηθάει αυτό ε, το θεματολόγιο μας. Παρακάτω τώρα. Όσον αφορά τις χώρες της ε, Αφρικής, βέβαια δεν μπορούμε να ε, κάνουμε γενικεύσεις. Όμως η δέσμευση των κυβερνήσεων είναι πολύ σημαντική. Περισσότερες χώρες έχουν θεσπίσει τις κατάλληλες πολιτικές. Αν κατά νου έχω τις κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες πρωθυπουργών και προέδρων η ισότητα αποτελεί μία από αυτές τις προτεραιότητες προέδρων, ε, πρωθυπουργών κλπ. Οπότε το θεματολόγιο έτσι βοηθάτε. Πολύ σημαντικό. Άλλο. Πολύ σημαντικό. Να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ σταθερότητας, ε, του πόσο ευάλωτη είναι κάποια κατάσταση ε, όσον αφορά την ισότητα. Μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα σε κάποιες χώρες. Αλλού όχι τόσο εύκολο. Όταν συζητούμε τις συστάσεις θα το ξαναπούμε αυτό. Επίσης έχουμε τους θρησκευτικού φορείς, τους παραδοσιακού φορείς, Πολλέ φορέ είναι προοδευτικοί αυτοί οι φορείς και θέλουν να προωθήσουν τα θέματα αυτά Αυτό το θεματολόγιο. Αλλού υπάρχει πολύ συντηρητισμός και αυτό είναι φραγμός. Επίσης οι σχέσεις των ε, δύο φίλων ε, είναι και συσχετισμοί ισχύω και δυνάμεων. Και οπότε αυτό επηρεάζει το τι πετυχαίνουμε βραχυπρόθεσμα. Για να δούμε τώρα τις προτάσεις, συστάσεις. Για μένα πολύ βασικό είναι να υπάρξει μια ανάταξη των προτεραιοτήτων. Δηλαδή οι γραφειοκρατίες προσπαθούν να τηρήσουν τις προτεραιότητες που τάσουν οι πολιτικοί. Πολλές φορές όμως οι πολιτικοί έχουν μια σειρά προτεραιοτήτων που δεν είναι ιεραρχημένες. Είναι για τους πολιτικούς όλες οι προτεραιότητες το ίδιο σημαντικές. Αυτό δυσκολεύει όμως ε, το προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, τους γραφειοκράτες να κάνουν κάτι. Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια. Θα πρέπει επομένως ε, οι τεχνοκράτες ας πούμε να έχουν σε κάθε στόχο ο πρόεδρο των πολιτικών. Αλλιώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό θα πρέπει οι πολιτικοί να έχουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την ισότητα. Θα πρέπει να τονιστεί πώ το θέμα τη ισότητα είναι πιο σημαντικό από άλλα θέματα τα οποία ε, απασχολούν τι ε, γραφειοκρατίε. Πώς αυτά επιβάλλονται, εισάγονται από έξω στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, έχουμε κάποια θέματα τέτοια τα οποία κρεμούν πολύ καιρό, οπότε θα πρέπει να γίνεται εξορθολογισμός των στόχων σε ορίζοντα βράχη πρόθεσμο και να βλέπουμε το πώς βήμα-βήμα μπορούμε τις διάφορες αλλαγές και ιδίως τις πολιτιστικές αλλαγές να τις καλύψουμε Αυτό πολλέ φορέ ε, αναδεικνύει στα θέματα διεθνού συνεργασία. Άρα θα πρέπει για κάθε χώρα να βοηθούμε, να δούμε και να λέμε το πόσο πρέπει να τα πράγματα. επίση, βοηθούν πάρα πολύ οι μα μας στη διαχείριση οι αντιπροσωπείες αυτές της χώρας. Ε, οπότε έτσι εκμεταλλευόμαστε τι τυχόν αναδυόμενε ευκαιρίε. Σε ένα και το καθημερινό σύστημα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολο όταν κάνει πρέπει να περιμένει πάντοτε από την κεντρική εξουσία επί πολλούς μήνες κάποια έγκριση πριν κάνει κάποια κίνηση. Τώρα, ε, ολοκληρώνοντας για τις ε, συστάσεις. Υπάρχει θέμα διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων ειδών αφρικανικών χωρών. Σε πολλές χώρες ε, υπάρχουν κάποιες κυβέρνησεις οι οποίες ε, ασχολούνται με ισότητα και χειραφέτηση. Ε, βοηθάν, βοηθάει η δημοσιονομική πολιτική, βοηθάει ο πολιτικό διάλογο, αλλά υπάρχουν και κάποιε κυβερνήσει που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα θέματα ισότητα. Εδώ είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και πρέπει κανεί να έχει στοχευμένε δραστηριότητε, όχι μέσω κυβέρνηση αλλά μέσω τη κοινωνία των πολιτών. Γιατί σε άλλε περιπτώσει που τα πράγματα είναι πολύ ευάλωτα, πολύ ευαίσθητα και εκεί χρειάζονται στοχευμένε δραστηριότητε σαν μέσο πολιτική. Τώρα τι γίνεται στις περιπτώσεις ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις. Εδώ θα πρέπει να δούμε ότι κάποιες προσπάθειες έχουν προηγηθεί, έχουν όμως αναστατωθεί, έχουν διακοπεί. Άρα μπορούμε να κάνουμε βήματα πρώτο μέσω πολιτικού διαλόγου και στοχευμένων δραστηριοτήτων. Και σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ δόκτορα Πέτρεσεν, τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Καπετάνοβιτς, ιατρό και βουλευτή της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Ε, μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Έχοντας κατά νου πως οι προτεραιότητες για το 2016-19 της ε, στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων βλέπουμε ότι η Κομισιόν επαναβεβαίωσε την δέσμευσή της για να προωθεί την ισότητα ανδρών και γυναικών. Θα σας υπενθυμίσω πέντε τομείς προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για να αυξηθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Δεύτερον, προώθηση τη ισότητα στην διαδικασία λήψη αποφασιών. Τρίτον, καταπολέμηση της ε, έμφυλη βίας. Τέταρτον, καταπολέμηση του χάσματος στην πληρωμή και στις συντάξεις. Και πέμπτον, βεβαίως, ε, τα Δυτικά Βαλκάνια. Μιλώντας για τα Δυτικά Βαλκάνια, οφείλω πρώτα απ' όλα να πω ότι οι νομικές διατάξεις σε γενικές γραμμές υπάρχουν. Η εφαρμογή τους βεβαίως είναι κάτι το διαφορετικό. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου της νομοθεσίας και των πολιτικών δεν εφαρμόζονται παρά το ότι προβλέπονται οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην δημόσια και την πολιτική ζωή. Μιλώντας για την για τις μόνιμες ε, επιτροπές ε, ισότητας των φύλων. Αυτές δεν έχουν συσταθεί στο επίπεδο της Ομοσπονδίας ε, λόγω της γνωστής κατάστασης με τα 10 καντόνια. Η έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας και της προστασίας από την έμφυλη βία και ειδικά την οικογενειακή βία παραμένει μια μεγάλη ανασυχία σοβαρή ανησυχία είναι και οι περιπτώσεις ε, βιασμών, ε, ακόμα και κοριτσιών, ακόμα και μέσα στην οικογένειά της και λοιπόν που το λέω και η παιδεραστή. Στατιστικά δεδομένα δεν υπάρχουν ακόμα για να μας ε, δώσουν μια εικόνα του πώς εφαρμόζεται ο νόμος. Ένα εναρμονισμένο σύστημα Παρακολούθηση συλλογή δεδομένων για την βία κατά των γυναικών ακόμα δεν υπάρχει. Η οικογενειακή βία δεν έχει ακόμα εναρμονισμένη νομοθεσία λόγω του περίπλοκου συνταγματικού ζητήματος. Και βεβαίως ε, υπάρχουν ε, και τα σχετικά ζητήματα και λυπούμε που το λέω και στην αστυνομία και στον δημόσιο τομέα. Η πρόσβαση σε... και αρρωγή και προσώπηση είναι πολύ χαμηλή και βεβαίως το γενικό σύστημα στήριξης των θυμάτων πρέπει να βελτιωθεί. Ε, ξενώνες ε, στις ε, περισσότερες περιπτώσεις υποχρηματοδοτούνται και παρά την υφιστάμενη νομοθεσία κάποιοι έκλεισαν ως αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης για την εκμετάλλευση των κοριτσιών και ακόμα και των παιδιών. Ε, δυστυχώς το φαινόμενο αυτό υπάρχει ακόμα στα Δυτικά Βαλκάνια, σε αυτό το οποίο λέμε Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα επίσης με τα άτομα με αναπηρία που περιλαμβάνουν και το ότι τα κρατικά επιδόματα είναι μικρά παρά την ύπαρξη ειδική υπηρεσία για τους αναπήρου και την στήριξη που λαμβάνουν ε, οι εργοδότες από το κράτος. Το κράτος, το Ομοσπονδιακό, δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα ε, για την απασχόληση γυναικών 40 ετών και άνω που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ηλικίας και φύλου. Επιπλέον, έχουν δοθεί επιδοτήσεις ε, στους νεαρούς και ειδικά στις νεαρές για την ε, πρώτη τους ε, είσοδο στην αγορά Αλλά ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αυξηθεί και η ευαισθησία του κοινού. Και βεβαίω θα πρέπει να σεβαστούμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να ενεργήσουμε κάθε μορφής διάκριση. Η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη ήταν μία από τις πρώτες χώρες που κύρωσε την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και εκπλήρωσε τους βιωσμούς στόχους ανάπτυξης 3 ε, έως 5. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία και ελπίζω να είμαστε ενωμένοι ισχυρότεροι στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Καπετάνοβιτς. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φελίν που είναι ανεξάρτητη ειδικό από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Ιταλίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για το εργαστήριο αυτό που συγκαλέσατε σήμερα. Πρώτα απ' όλα να σας συστηθώ. Φέλη, είναι... εργάζομαι στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της ε, Ρώμης ε, και βεβαίω ανήκω και στο δίκτυο γυναικών που εργάζονται στην διεθνή ασφάλεια. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το θέμα, το οποίο είναι ευρύτατο, αλλά λόγω της εμπειρίας μου αποφάσισα να ασχοληθώ στον θεματικό πυλώνα ΔΕΛΤΑ για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και τη συμμετοχή κορίτσιων και γυναικονία που είμαι ειδική για την ασφάλεια του φίλου. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το περτίνος ακριβώς Η δουλειά μου εστιάζει κυρίως στο ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ και τα σχετικά και βεβαίω το περιβάλλον ασφαλείας έχει αλλάξει και βλέπουμε πως υπάρχουν πλέον προκλήσεις ασφαλείας. Είναι δύσκολο να αναφερθούμε στα ζητήματα ισότητας ε, χωρίς ε, να δούμε το τι θα γίνει με την ευθύνη για τις γυναίκες στην διάρκεια των συγκρούσεων. Επρόκειτο λοιπόν για ένα ψήφισμα το οποίο θετήθηκε το 2000 μετά από έναν αγώνα των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών που πάλευαν για δύο και η ευθύνη των γυναικών στα θέματα ασφαλείας. Μέχρι τότε αυτό ήταν ένα από τα λεγόμενα ήπια ζητήματα και υπήρχε λοιπόν μια αλλαγή για το πώς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ αντιμετωπίζει το ζήτημα. Θα αναφερθώ λοιπόν στην εφαρμογή του 1325 που εστιάζει στην Αφρικανική Ήπειρο. Όταν μιλάμε λοιπόν για ζητήματα φίλου βλέπουμε πάντοτε υπάρχει μια διαφορά μεταξύ συμμετοχής ε, και προστασίας. Το ανέφερε και η πρέσβυρα, κυρία Μαρινάκη, και αναφέρθηκε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Νέα Υόρκη. Είναι δύσκολο λοιπόν να φέρουμε το ένα και όχι το άλλο και κανείς δεν μπορεί να πει ότι το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Πρέπει να το δούμε όλα λοιπόν, αλλά αν δεν έχουμε ε, ένεργο συμμετοχή των γυναικών είναι και δύσκολο να είναι πιο προστατευμένες ε, και στα... στον χώρο του σπιτιού. Έχουμε λοιπόν τις βασικές αρχές που υπάρχουν στο ψήφισμα 1325 το οποίο βασίζεται στην πρόληψη, συμμετοχή και προστασία και περιλαμβάνει ακριβώς και την ένταξη της διάστασης του φύλου. Πέρσι λοιπόν υπήρξε μια μετατόπιση στο αφήγημα και περάσαμε περισσότερο στην συμμετοχή και την προστασία. Τώρα έχουμε βρει μια ισορροπία για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν λοιπόν, στη Νέα Υόρκη σε αρκετές εκδηλώσεις για την σημασία συμπερίληψης των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων. Και βεβαίως αυτή είναι μία από τις πτυχές που επίσης περιλαμβάνεται στο θέμα αυτό. Οι τέσσερις στόχοι λοιπόν είχαν ήδη αναφερθεί για την πυλώνα Δέλτα που είναι βεβαίως κάτι το πολύ ισορροπημένο γιατί έχουμε ήδη κάποιους πυλώνες που αφορούν την προστασία και έναν πυλώνα που αφορά την συμμετοχή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ποια είναι η γενικότερη τάση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καλή εφαρμογή της έκθεσης ε, στο σύνολο της αντιπροσωπείας όπως είχε παρουσιαστεί αλλά οφείλω να πω ότι όταν ερχόμαστε στο συγκεκριμένο τομέα υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Από τη μία βλέπουμε στο πολιτικό επίπεδο έχουν γίνει πολλά και με τον διορισμό του 2015 συμβούλου για το φύλλο που εστιάζει στα θέματα των γυναικών της ασφάλειας και της ειρήνης την ε, πρέσβερα, την κυρία Μαρινάκη δηλαδή έχουμε και την άτυπη task force που συνεδριάζει τακτικά αλλά όταν περνάμε στην αντιπροσωπεία βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη εφαρμογής και Βεβαίω η έκθεση λέει ότι ο στόχος 17 που μιλάμε για ίσα δικαιώματα και συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα ήταν ένα στόχος που επέλεγαν περισσότερο οι αντιπροσωπείες 53 από τις 111 αλλά μετά όταν περνάμε συγκεκριμένα στην εφαρμογή του σχεδίου στην υποσαχάρη Αφρική και στις μεγάλες λίμνες ε, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου εφαρμογή. Ε, υπήρχαν δύο έργα, ένα πιο γενικό στην Αιθιοπία που αφορούσε την ισότητα και τη συμμετοχή των γυναικών και ένα άλλο στην Ιγυρία το οποίο θεωρούσαμε μια βέλτιστη πρακτική, ένα πολυετές σχέδιο που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, επιτόπου υλοποιεί η UNICEF και η UN Women για τον ρόλο των γυναικών στον τομέα της ασφαλείας και την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων δράσης. Και όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά η στήριξη της εφαρμογής σε τρεις διαφορετικές περιφέρειες. Οπότε, εγώ προτείνω να δούμε πώς μπορεί να επαναληφθεί και να προσαρμοστεί βεβαίως το σχέδιο αυτό και σε άλλες χώρες. Και στα διδάγματα που αντλήσαμε και τις συστάσεις, ε, πολλά από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί, έχουμε ένα πολύ σωστό κένο, μια πολύ καλή δομή, με συγχωρείτε, καλύτερη από το παρελθόν και έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση, ειδικά στο επίπεδο των κεντρικών γραφείων και της αντιπροσωπείας. Πάντα λοιπόν πρέπει να ηγούμαστε δια του παραδείγματος και ειδικά στα ζητήματα ισότητας γυναικών και ασφάλειας όπου συχνά έχουμε πολίτες και στρατιώτες να συνεργάζονται στενά. Έχουμε πιο μόνο αποτελέσματα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πιο συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της ισότητας. Δεν ξέρουν όλοι οι ειδικοί της ισότητας αυτήν την ατζέντα, ούτε είναι μαθημένοι να συνεργάζονται με στρατιωτικούς, οπότε καλό θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία όταν πηγαίνουμε σε περιοχές με συγκρούσεις. Οπότε είναι σημαντικά αυτά να μην υπάρχει μόνο ένας ειδικό για το φύλλο, αλλά και η εμπειρία που θα περιλαμβάνει βεβαίως ε, και τη γεωγραφική και θεματική διάσταση και όχι μόνο τη διάσταση του φίλου. Αυτά τα έχουμε βεβαίως, ε, υποστηρίζονται από το έργο των αντιπροσωπιών και όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, λίγες αντιπροσωπίες κάνουν συγκεκριμένη αναφορά. Επίσης ε, βλέπουμε ότι ε, πρέπει να κάνουμε και περισσότερα πράγματα για τους άντρες και τα αγόρια. Μιλάμε για τις γυναίκες, αλλά ε, η κοινωνία αποτελείται και από άντρες. Οπότε δύσκολα μπορούμε να σκεφτούμε θα προωθήσουμε τις γυναίκες όταν την εξουσία έχουν οι άνδρες, αν δεν εργαστούμε για μια συνολική αλλαγή. Και όταν μιλάμε για συγκρούσεις είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μια άλλη πτυχή που δεν αναφέρεται στην έκθεση είναι τα ΜΜΕ και το πώς αναφέρουν τις συγκρούσεις. Οπότε πρόοδο σε αυτό το μέτωπο είναι πολύ σημαντική και ως μια γενική συζήτηση, όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν μπορούμε να λέμε Αφρική γενικώ, πρέπει να προσαρμόζουμε τα έργα αναλόγως με την κατάσταση. Λογικό αυτό. Όταν μιλάμε τώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή τη στιγμή θεωρώ πως θα μπορούσε να ενθαρρύνει την έγκριση ενός ψηφίσματος για τις χώρες αυτές και για την πτυχή της μεσολάβησης. Η Αφρικανική Ένωση εργάζεται πάρα πολύ στο θέμα αυτό και στα δικτύα γυναικών μεσολαβητών και σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πιο γεωγραφικό για να εστιαστούμε περισσότερο στο θέμα αυτό Ίσως και να προτείνουμε μια σοβαρότερη ανάλυση στην εφαρμογή της 1835 ε, και βέβαια όταν υπάρχουν και ανταλλαγές ε, βουλευτών να εξετάζουμε αν υπάρχει π.χ. ισορροπία του φύλου και σε ποιο βαθμό η Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει το 1325. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, η σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φελίν για την παρουσίαση. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Νόρα Ζαμπέρ. ερευνήτρια του King's College του Λονδίνου. Εγώ θέλω να μιλήσω για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Δράσης στην Αραβική Χερσόνησο, η οποία αποτελείται από την Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Παχρέιν, τα Ηνωμένα Εμμυράτα, Ιράκ και η Εμένη. Πάλι δηλαδή εδώ τίθεται θέμα γενικο... γενίκευσης μάλλον, δεν μπορεί κανεί να γενικεύει, οπότε δεν θα τα ξαναπώ. Έχω τρία ζητήματα που νομίζω ότι καλό να τα σκέπτεται κανείς όταν αναλογίζεται πώς θα εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Δράσης. Το βασικό είναι η πλαισίωση από άψη πολιτισμική λόγω των διαφόρων πολιτιστικών πλαισίων είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια τοπική προσέγγιση για την ε, εφαρμογή της GAP. Δηλαδή μπορεί αυτή μένα να είναι παγκόσμια, αλλά ο τρόπος που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή πρέπει να ληφθεί υπόψη το Ισλάμ, με άλλα λόγια. Και το σχέδιο GAP να γίνει συμβατό με το Ισλάμ, διότι ανεξαρτήτως του τι σκεπτόμαστε εδώ δεν είναι μονάχα διακυβερνητική υπόθεση. Μελέτε έχουν δείξει ότι και το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού σε ολόκληρη την περιοχή το βρίσκει πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το Ισλάμ ω στοιχείο της ταυτότητάς του. Πρέπει να παρουσιαστεί λοιπόν η GAP με κάποιο τρόπο που να είναι συμβατό με το Ισλάμ. Θα είναι λοιπόν ευκολότερο τότε να το αποδεχτεί ο τοπικό πληθυσμό κάνει και τις κυβερνήσεις να είναι λιγότερο, να ανθίστανται λιγότερο στο GDP, αλλά βέβαια και τον κόσμο. Πρέπει να ερμηνευτεί το Ισλάμ με κάποιο, κάπως προοδευτικότερο τρόπο και λιγότερο αποκλειστικό για τις γυναίκες. Υπάρχουν και πολλοί μελετητές του Ισλάμ που έχουν πει σχετικά πράγματα και είναι ε, σωστό να έρθει κανείς σε επαφή με τους ε, στοχαστές αυτούς του Ισλάμ και τους μελετητές του Ισλάμ για να δει πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα πράγματα αυτά αυτό ίσως μπορεί να προωθηθεί ασφενώ μέσω τη εκπαίδευση αφετέρου μέσω των κοινωνικών μέσων. Γιατί και, και στα κοινωνικά μέσα όλος ο κόσμος έχει πρόσβαση εκεί. 80% του πληθυσμού εκεί στις χώρε αυτές έχει πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα και μάλιστα είναι και πολύ δραστήριος. Το σχέδιο πρέπει να ενταχθεί και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθηση τη ισότητα των φύλων. Οι περισσότερες κυβερνήσεις της Αραβική Χερσονήσου έχουν κυρώσει τον χάρτη για την αποφυγή διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Αντί λοιπόν να παρουσιάσει κανείς το GEP σαν κάτι το καινούριο, το απολύτως νέο, ίσως σωστό είναι να τονιστούν οι ομοιότητες μεταξύ διεθνών εγγράφων, διεθνών ε, ψηφισμάτων που έχουν ήδη υιοθετηθεί και το τι μπορεί να γίνει επιτόπου στην περιοχή και ο κόσμο πρέπει να αντιληφθεί καλύτερα τι είναι το GAP. Εγώ προέρχομαι από την περιοχή αυτή και δεν νομίζω ότι όλο ο κόσμο γνωρίζει. Δεν γνωρίζουν καν οι άνθρωποι εκεί ποια δικαιώματα κατοχυρώνονται στα συντάγματά του. Αυτά μπορούν να γίνουν ε, με μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή και των τοπικών οργανώσεων τη ε, κοινωνία. Κυβερνήσει και κοινωνία των πολιτών δεν εργάζονται με τον ίδιο τρόπο όπω εδώ για παράδειγμα ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Αντί λοιπόν να οργανώνονται ομάδες γυναικών, οι άνθρωποι εκεί βρούν περισσότερο ατομικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να καθορίσουμε ποιοι θα είναι οι φορείς που θα συμβάλλουν. Συχνά μπορεί να είναι μελετητές, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, και αντί να βγαίνουν στους δρόμους οι άνθρωποι αυτοί δρούν περισσότερο μέσω των γραπτών τους. Κάτι άλλο είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτό μπορεί να ενσωματωθεί και στην εκπαίδευση. Διότι πρέπει να μπει σε μια μεγαλύτερη, σε μια ευρύτερη προσπάθεια να αλλάξουν οι κοινωνικοί κανόνες, οι νόρμες. Και μέσα από, αυτό, από αυτούς τους διάβλους λοιπόν να μπορέσει να περάσει η προσπάθεια για την πρόθεση της GAP. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κυρία Ζάβερ. Τώρα, θα δώσω τον λόγο σε όποιον το επιθυμεί, δηλαδή στους ε, ευρωβουλευτές πρώτα. Πρώτος εσείς κύριος Γκέρικε, κύριε Γκέρικε, συγγνώμη. Εσείς κύριε Γκέρικε, ορίστε. Εγώ εργάζομαι στην Ισομερή Συνέλευση των χωρών ΑΚΕ, από τις οποίες 46 είναι Αφρικανικέ Οι χώρες δηλαδή Αφρική Καραϊβική, Ειρηνικού. Αν με επιτρέψετε όμω να αλλάξω τη γλώσσα και να μιλήσω γερμανικά που αισθάνομαι ασφαλέστερο. Συζητούμε συχνά ότι τα διάφορα project συνδέονται με όρους και εκεί μιλεί κανείς συχνά και ε, πολύ για το φύλλο. Μιλούμε για gender equality και μιλούμε και για women empowerment. Τι, μιλούμε, τι εννοούμε gender όταν μιλούμε για gender equality. Μιλούμε για ε, πτυχές του φύλου. Μιλούμε για ανισότητα των φύλων, μιλούμε για χάσμα μεταξύ των φύλων. Και συχνά βλέπω εδώ ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε διάφορα έργα στην Αφρική, εμφανίζονται πλέον δύσπιστοι και δεν είναι διατεθειμένοι να καταπιούν οτιδήποτε, αλλά θέλουν να ελέγξουν, θέλουν να ελέγχουν τι εννοούμε όταν μιλούμε για ισότητα φύλων. Τι σημαίνει η έννοια φύλο, gender, διότι καμιά φορά προκαλεί παρανοήσεις η χρήση του όρου αυτού, ακόμα και στη δική μας την Επιτροπή. Παρόλο που μιλούμε δηλαδή για ισότητα και θέλουμε να επιτύχουμε κάτι το θετικό, ωστόσο είναι σημαντικό να μπορούμε να εξηγήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αναγκαίο ότι γνωρίζουν όλα τα κοινοβουλευτικά, τι ακριβώς εννοούμε. Ευχαριστώ κύριε Γκέρικε, λέει η πρόεδρο. Άλλο κανείς ε, δεν υπάρχει ή να θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση ή να θέσει κάποια ερώτηση. Να παρακαλέσω λοιπόν τις εμπειρογνώμονες και του εμπειρογνώμονες, ποιο θα ήθελε να απαντήσει στον κύριο Γκέρικε, στο σχόλιο του κύριου Γκέρικε. Θέλετε εσεί κύριε Αφελίν. Ορίστε παρακαλώ. Ναι, γι' αυτό Μίλησα και για την ανάγκη να συμπεριλάβουμε και τους άντρες και τα αγόρια, τους, νέους, τους νεαρούς δηλαδή. Gender δεν σημαίνει μόνο τις γυναίκες. Αλλά το πώς έχει φτιάξει τους ρόλους η κοινωνία των ανδρών και των γυναικών. Όταν θέλουμε να απλουστεύσουμε, χρησιμοποιούμε απλούς όρους όπως το άρεν φύλλο και το φίλοι φίλο, γιατί δεν έχουμε και τον χρόνο να βάλουμε μέσα και ε, τις διάφορες ε, αποχρώσεις ε, των ε, ομοφιλοφιλικών τάσεων κλπ. Επειδή λοιπόν οι γυναίκες παίζουν και διαφορετικούς ρόλους μέσα στην κοινωνία, θέλουμε να προσφερθούν στις γυναίκες οι ίδιες ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες στη ζωή. ίδιο και ευθύνες. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο σε περιπτώσεις συγκρούσεων, ιδίως λόγω του παραδοσιακού του ρόλου. Αυτό δηλαδή που εμείς αμφισβητούμε είναι ακριβώς αυτό. Θέλουμε να τους προσφερθεί η ευκαιρία να παίξουν ενεργούς ρόλους και να αλλάξουν πλέον τα καθιερωμένα σχήματα. Θέλουμε βέβαια ίσες ευκαιρίες, αλλά μέσα στα πλαίσια του σεβασμού της ποικιλότητα των διαφορετικών δύσκολο να εξηγηθεί, γιατί συχνά άνθρωποι οι οποίοι αγνούν τα πράγματα αυτά, έστω και καλή την πίστη, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνουν τα πράγματα αυτά. Και εγώ όταν κάνω εκπαιδεύσεις και κάνω εκπαιδεύσεις ε, σε ομάδες που θα αναλάβουν ειρηνευτικό ρόλο, οι άνθρωποι αυτοί συχνά ε, είναι διστακτικοί σε ό,τι αφορά την ε, ισότητα των φίλων. Ξεκινώ από την υπόθεση ότι όλοι είμαστε υπέρ της ισότητας των φίλων. Δεν θέλουμε όμως να καταργήσουμε τις διαφορές. Θέλουμε να τονίσουμε τις διαφορές και τις διαφορετικές πτυχές, αλλά και τη διαφορετική συνεισφορά που προσφέρουν γυναίκες, άνδρες, ε, νέα κορίτσια, νέα αγόρια στην ε, κοινωνία. Και όσοι εργάζονται στην αντιπροσωπή αυτή ε, τα γνωρίζουν τα πράγματα αυτά. Και γι' αυτό χρειάζεται εκπαίδευση σε ισότητα ευκαιριών και ισότητα φύλων για όλου όσου συμμετέχουν. Και το μήνυμα πρέπει να περάσει με τον σωστό τρόπο. Ευχαριστώ κυρία Φελίν. Να προσθέσω κάτι, λέει ο κύριος Γκέρικε. Ναι, βεβαίω. Όταν μιλούμε για ίσα δικαιώματα των φίλων, σωστό αυτό, είναι θετικό και ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω βέβαια γιατί ξέχασα να το κάνω πριν ε, ε, για το έργο που επιτελείται είτε στον Αφρικανικό χώρο είτε και παγκοσμίω. Ε, όπου κανείς πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλές ευαισθησίες. Τώρα, όταν κοιτώ στο Facebook, και για αυτό το πρόβλημα μιλάμε τώρα, βλέπω μέχρι και 60 και 70 διαφορετικές πτυχές φύλου ή gender. Αυτό όμως συγχαίει τον κάθε Αφρικανό που δεν μπορεί να κατανοήσει τι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν η Κομισιόν μιλεί για gender equality, μιλεί για ισότητα ή συμμεταχείριση ανδρών και γυναικών. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω με εδώ. Και αυτό θέλω να προτάξω. Και μετά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που κάνετε και θέλω να πω και μπράβο σας και ελπίζω να συνεχιστεί η εργασία σας αυτή με αυτόν τον τρόπο. Dr. Lars Engert Πέντερσεν, ορίστε εσείς παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κατανοώ την έκκλησή σας για να υπάρξει κάποια σαφήνεια σε αυτό το gender equality, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρη σαφήνεια. Έκανα μια σε βάθος μελέτη της δανέζικης στρατηγικής στον τομέα του gender equality και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές νοοτροπίες, τρεις διαφορετικές ερμηνείες του gender equality στα στρατηγική αυτή. Πολύ συχνά σε διαφορετικά πλαίσια θα δείτε διαφορετικές κατανοήσεις για το τι σημαίνουν τα πράγματα αυτά και δεν μπορούμε να πούμε άπαξ και διαπαντός αυτό είναι. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις διαφορετικές καταστάσεις και αυτό ε, έτσι κατανόησα πριν αυτό που είπατε Νόρα ότι δηλαδή πρέπει να πάρουμε την ατζέντα αυτή και να την προσαρμόσουμε στο διαφορετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Αλλά να μην ξεχνούμε τον βασικό στόχο ότι αγωνιζόμαστε κατά των διακρίσεων και κατά της περιθωριοποίησης ορισμένων ατόμων λόγω του φίλου τους, όποιο και είναι το φίλο αυτό. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ακόμη. Οι Δανείοι μιλούν για τις ίσες, ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες. Όλο αυτό λένε, ίσες, ίσες, ίσες. Βλέπω έξω μάλιστα μία αφίσα για μία έκθεση της Σιμών Βέη και σε ε, μία από τις φράσεις που παραθέτουν έξω είναι ότι ένα από τα πράγματα που θα ήθελε να δει θα ήθελε να μην την βάλουν σε μοντέλο αρσενικού ρόλου αυτό λέει η gender equality πρέπει να ανοίγει χώρο και για διαφορετικά φύλλα και για διαφορετικές τάσεις ή διαστάσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα πρόκειται για προστασία των διαφορών και να δοθεί χώρος και στις διαφορές. Βασικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε μια και καλή άποψη για να καθορίσουμε τι σημαίνει gender equality για όλες τις περιστάσεις. Η κυρία Οχουσμένοβα Ευχαριστώ. Ερώτηση για την κυρία Ζάμπερ. Αγαπητή Νόρα, μετά από την παρούσα ακρόαση, ποιες είναι οι προσδοκίες σας. Τι θεωρείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να φανούν χρήσιμα, μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι μουσουλμάνες, οι μουσουλμάνες γυναίκες στον αραβικό κόσμο να μπορέσουν να είναι πιο θαραλέες, πιο δραστήριες, ώστε η ισότητα μεταξύ των φίλων να υλοποιηθεί. Δεν προσδοκάτε από την ε, αφράση. Ευχαριστώ. Ορίστε κυρία ε, Ζάμπερ. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνάς μου στρέφεται γύρω από τον ρόλο του διεθνούς δικαίου και ιδίω για να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών των φίλων δηλαδή στην Σαουδική Αραβία πιο συγκεκριμένα. Και βλέπω ότι δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Είμαι λοιπόν λίγο απεσιόδοξη, για να είμαι ειλικρινή δηλαδή. Και ο βασικό λόγο είναι ότι δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν του στόχου αυτού και τα δικαιώματα που έχουν. Για να γίνουν αποτελεσματικά τα πράγματα αυτά πρέπει να προωθηθούν με τέτοιο τρόπο που οι άνθρωποι και να τα κατανοήσουν και να τα δεχτούν. Αυτό σημαίνει προσαρμογή στη γλώσσα και προσαρμογή στα πολιτιστικά δεδομένα των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να πάμε από εδώ και να πούμε στον κόσμο εκεί τι να κάνει και πώς. Θέλουμε, αυτό που θέλουμε είναι να τα, τα δουν και να τους ρωτήσουμε μετά πώς τα αισθάνονται. Οι περισσότερες γυναίκες στη Σαουδική Αραβία δεν θέλουν μεγάλες αλλαγές. Στατιστικά αυτό είναι και θεμελιωμένο, τεκμηριωμένο. Πρέπει όμως να δοθεί ευκαιρία στις γυναίκες που θέλουν να αλλάξει κάτι, να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Και αν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή, θα πρέπει να προέλθει από κάπου που να μπορούν να κατανοήσουν. Και πιθανότατα από κάποια θρησκευτική διάσταση και από κάποια θεμελιωμένη πολιτιστική διάσταση. Μέχρι ότου σημείο αυτό και δεν το έχω δει να συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο ακόμα. Αν λοιπόν δεν συμβεί αυτό, δεν νομίζω να αλλάξουν πολύ τα πράγματα, διότι πρόκειται για ισχυρότατε κυβερνήσει οι οποίε ε, κυβερνούν με πυγμή και κανεί, όλο ο φοβάται να τι προκαλέσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν ήμουν παρούσα από την αρχή, αλλά θέλω να διευκρινίσω ένα πράγμα. Διότι στην ομιλία του κ. ζωή να μην φάνηκε καθαρά ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω πλειοψηφία έχει η γνώμη ότι οι Αφρικανίδε και οι Αφρικανοί έχουν ακριβώ τι ίδιε δυνατότητε να αντιληφθούν διανοητικά περίπλοκα πράγματα. Και γι' αυτό η κάπω ρατσιστική δήλωση ότι οι Αφρικανοί ορισμένα πράγματα δεν τα κατανοούν για μένα είναι πάρα πολύ προβληματική. Βιολογικά, μάλιστα, υπάρχουν και παραπάνω από δύο φύλλα και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και στη φεμινιστική ε, εργασία μας και στην εργασία με ε, γυναίκες και νεαρά κορίτσια. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντκε. Σχόλια. Η κυρία Φέλιν. Ίσως να μην εκφράστηκα σωστά ότι δεν πρέπει να προστατεύσουμε. Ναι, ναι, κατάλαβα τι είπατε, κατάλαβα τι είπατε. Συμφωνώ μαζί σας. και στο εκπαιδευτικό υλικό ίσως πρέπει να το εντάξουμε αυτό καλύτερα, δηλαδή την διαφοροποίηση των φύλων. Διότι και αυτά που διαβάζει κανείς στις διεθνείς δημοσίευσεις αναφέρονται συνήθως σε δύο φύλλα. Όπως είπα λοιπόν πρέπει να δώσουμε περισσότερο χώρο και να επικαιροποιήσουμε και το υλικό μας και βεβαίως και τι προωθούμε και τη γλώσσα αυτών των πραγμάτων που προωθούμε. Μάλιστα. Δύο λεπτά για τελικά σχόλια των εμπειρογνωμόνων μας. Θέλετε εσείς να πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι για αυτή την θεσμική πολιτική μετακίνηση. Είναι τολμηρό και θαραλέο από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που κάνουν την προσπάθεια αυτή. Όμω είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν είμαι βέβαιος ότι πέραν του leadership commitment τα υπόλοιπα θα αποδώσουν. Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα πράγματα και νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη ουσιοδός ουσιώδους μάλλον αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών διότι και πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν από το προσωπικό διότι υπάρχουν και τεράστια οργανωτικά θέματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Με την έννοια αυτή δεν αρκεί να προσπαθήσει κανείς να πει ότι χρειάζεται καλύτερη παρακολούθηση, καλύτερη αξιολόγηση, ε, να διαθέσουμε τους αναγκαίους πόρους κλπ. Πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες, την καθημερινή εργασία, την καθημερινή εργασιακή επιβάρυνση του προσωπικού. Και αυτό σημαίνει ότι η πολιτική με τη σειρά σα πρέπει να θέσετε, να θεσπίσετε λιγότερε προτεραιότητε. Λοιπόν, πολύ το λέω αυτό. Οι προτεραιότητε που θα ε, θεσπίσετε πρέπει να είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Αν θέλετε η policy ατζέντα να προχωρήσει, αφήστε τι άλλε προτεραιότητε. Αυτό όμω ίσω να είναι και δύσκολο για σας. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ. Η κυρία Μαρινάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προχωρώ το επιχείρημα κάπως περισσότερο. Από τη δική μας πλευρά ως Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός, ε, το, το gender mainstreaming είναι κάτι το οποίο τέμνει όλες τις πολιτικές μας θεματικά καθώς και γεωγραφικά στο πλαίσιο της ένταξης των στοιχείων του φύλου στις συζητήσεις, αυτό θα πρέπει να γίνει ρουτίνα και όχι εξαίρεση. Έως τώρα, από πέρσι, και αυτό απηχήθηκε επίσης στην έκθεση του Gender Action Plan, έχουμε περιλάβει ζητήματα γυναικών, φίλων και ειρήνης σε όλους τους διαλόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 41 διαλόγων που έγιναν πέρσι σε υποεπιτροπές, πολιτικές συζητήσεις κλπ. έχουν πάντοτε τέτοιο στοιχείο, στάνταρτ. Και αυτό είναι ένα βήμα μπροστά, διότι δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να εντάξουμε τα στοιχεία που έχουν σχέση με την γλώσσα που χρησιμοποιούμε ως ένα στοιχείο, ένα στάνταρτ στοιχείο για τους πολιτικούς ηγέτες μας. Δηλαδή να μπει παντού και στις διασκέψεις κορυφής, στον πολιτικό διάλογο, οι ηγέτες μας να μεταδώσουν το μήνυμα με τρόπο που να περάσει πραγματικά, όπως ήδη εξήγησε ο δόκτωρ Πέτερσεν, μέσα σε αυτή την ε, θεσμική πολιτιστική ε, μετατόπιση, διότι τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει δεν φτιάχτηκαν σε μία μέρα, ούτε θα φύγουν σε μία μέρα ή ένα χρόνο. Είναι μακροχρόνια διαδικασία και προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα αυτά. Δεν πρόκειται για ταχεία κίνηση. Ευχαριστώ κυρία Πρέσβυρα. Ε, άλλα σχόλια δεν υπάρχουν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τα όσα είχα την ευκαιρία να ακούσω. Πολύ υποστήριξη δηλαδή. Και οι αναλύσεις των εμπειρογνωμόνων κινούνται άλλωστε προς την ίδια κατεύθυνση και αποτελούν οδηγό για μας. Και πολύ σημαντικό αυτό, διότι είπε και κάποιος ότι είμαστε ένα, μια ομάδα λίγων ανθρώπων μέσα σε μια μονάδα προσπαθούμε να προωθήσουμε τα πράγματα αυτά. Είμαστε όμως, τα καταφέρνουμε όμως καλά και γι' αυτό χρειάζεται ηγεσία. Συμφωνώ ότι δεν αρκεί. Δεν αρκεί ο Επίτροπος ή η Επίτροπος ή ο Γενικός Διευθυντής για να επιφέρουν την αλλαγή. Προδιετίας είχαμε συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής τη συνεργασία, όλων των επικεφαλή συνεργασία για την εφαρμογή του χάρτη σε μια αίθουσα όπως περίπου τούτη εδώ. Μπροστά μου κάθονταν όλοι αυτοί. Ήταν 12 η ώρα, το ζήτημα του gender equality ήταν στην ημερήσια διάταξη. Δύο πράγματα παρατήρησα ενδιαφέροντα και ίσω ορισμένοι να τα έχετε ακούσει. Το ένα είναι 80% ε, των προσώπων που κάθονταν μέσα ήταν άνδρες. Γιατί, Γιατί πρόκειται για θέσεις ιεραρχικά ανώτερες γιατί χρειάζεται χρόνος και να έχει ε, καλυφθεί μεγάλη πορεία στη σταδιοδρομία, άρα εκεί καταβάλλεται κάποιο τίμημα για την έλλειψη αυτή αντιπροσώπευσης. σαν ήσταν μιλώ, 20-25 από τους συναδέλφους μου σηκώθηκαν πάνω και έφυγαν. Απεχώρησαν από την αίθουσα. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η πολιτιστική θεσμική μετατόπιση όταν μου λέει η υπηρεσία μου ότι πρέπει να τα κάνει τα πράγματα αυτά, σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θα τα κάνουν πρέπει να είναι και πεπισμένοι. Από την άλλη μεριά κάθονται μαζί μου εξαιρετικά ικανοί συναδελφοί οι οποίοι έχουν καταδείξει πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα τα θέματα του φίλου στις χώρες όπου ε, ασχολούνται και, και σε γλώσσα που κατανοούν και οι άντρες. Αλλά πρόκειται για μαραθώνιο και μια και στη Ελληνίδα, η κυρία Μαρινά Κενό, γνωρίζει πολύ καλά τι είναι ο μαραθώνιος δρόμος και δεν θα αλλάξει το χρόνο, θα χρειαστεί πολλή χρόνος. Αυτό που είναι ενθαρρυντικό από τη δική μου πλευρά είναι ότι μπαίνει μια νέα γενναία στα πράγματα ως συνάδελφοι στις αντιπροσωπείες και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, επιφέρει μεγάλη διαφορά. Α, αμέσως αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά των αντιλήψεων. Πώς δηλαδή κατανοούν και πώς θεωρούν σημαντικά τα θέματα των φίλων. Δεν ε, ασκώ καμία κριτική, ε, απλώς περιγράφω τα πράγματα και πώς θεωρώ ότι θα εξελιχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Ρίλε. Δεν έχω άλλα σχόλια. Η κυρία Ντομπράβκα Σουίτσα μέσω μηνύματος που μας απέστειλε ε, με βίντεο. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα θα ήθελα να σα ζητήσω συγγνώμη που είμαι απούσα. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλες και όλου του συναδέλφου. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία τόσο ώστε να μπορέσουμε να προαγάγουμε την υπόθεση ζωή των δύο φίλων όπω επίση και να προστατεύσουμε τι γυναίκε και τι νεαρές γυναίκε όσον αφορά τα δικαιώματά του και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτε χώρε, Μετά από τόσε δεκαετίε προσπαθειών η απόσταση και αυτό το χάσμα ε, δικαιωμάτων των και γυναικών παραμένει μεγάλο. Η κυρία Μακάβαν και οι υποφαινόμενοι συναντήσαμε τους πρέσβες από Βοσνία ε, Κονγκό, Σενεγάλη και έτσι είχαμε μια βοήθεια για να δούμε το ευρύτερο τοπίο. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης ε, υπαριθμών 2 που μας δείχνει ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την ισότητα των ε, φίλων. Εάν μπορέσουμε αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσουμε πλήρως πρόκειται να αυξήσουμε τις ευκαιρίες για γυναίκες και νεαρές κοπέλες να βελτιώσουν τις ζωές τους και να μπορέσουν να απολαύουν των δικαιωμάτων που έχουν και πρέπει να σβήσουμε τις ανισότητες για να πετύχουμε ειρήνη, ανάπτυξη. Είναι μεγάλη μου χαρά το ότι είμαι συνεισηγήτρια για αυτό το σημαντικό θέμα. Συνεργαζόμαστε αγαστά με την κυρία Μακάβαν. Ε, τα πράγματα φαίνεται ότι θα πάνε καλά και είμαι σίγουρη θα βρούμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας και όλοι θα δώσουμε αυτή τη μάχη για την ισότητα των φίλων. Σα Σας ευχαριστούμε, κυρία Σουίτσα. Και τώρα ο κύριος Πονγκά πρόκειται να κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μπλινκεβιτσούντε. Πρόεδρε της Επιτροπής ε, Θεμάτων των Γυναικών. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι των δύο επιτροπών, σας ε, ευχαριστώ για την ανταλλαγή αυτών των απόψεων που ήταν τόσο παραγωγική. Και ελπίζω ότι το καινούργιο πρόγραμμα δράσης για την ισότητα των φίλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρόκειται να μας ε, επιτρέψει να αναδείξουμε το θέμα της χειραφέτησης γυναικών και νεαρών γυναικών σε όλο τον κόσμο. Οπότε να υπάρξει μια συνένεση ούτω ώστε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε ευθύνε, ότι είναι καθήκον μα προ τι υπερχόμενες γενναίε. Πρόκειται για κάποια αλλαγή κουλτούρα, αλλαγή θεσμική που επιτελείται και χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε το θέμα τη ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι μόνο κάποια πάγια ρήτρα που θα πρέπει να τηρείται σε κάθε πρόγραμμα με τις ε, χώρες εταίρους. Πρόκειται για κάποια δέσμευση που θα πρέπει να υπάρξει σε κάθε επίπεδο όσον αφορά την εξωτερική μας δράση, απλώς πολιτική πολιτικής και διπλωματικής, αλλά ε, και ε, οικονομικής. Οπότε θα πρέπει να σας τονίσω ακριβώς όπως προβλέπει το πρόγραμμα δράσης ότι οι άνδρες και αυτοί οφείλουν να επιτελέσουν το ρόλο τους ούτως ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα θα πρέπει να αρθούν όλες αυτές οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών αγαπητοί συνάδελφοι. Επομένω εδώ κηρύσω ε, την ε, λήξη του, κοινή μα μας ε, συνάντησης, την ε, λήξη σε αυτό το εργαστήρι και η συνάδελφοι της Επιτροπής Ανάπτυξης σας έρθουν μαζί μου. Ας ε, έρθουν μαζί μου λέγω στο απέναντι κτίριο στην αίθουσα 4β, το κτίριο PH Εσ. Η κυρία Μπλυνκεβιτσούτε, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Thank you very much.